Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι και το τελευταίο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Είναι η έκθεση Ντελάνγκε, μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Ντελάνγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω βεβαίως ε, Ολλανδικά. Ε, και εμένα, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ούτως ή άλλως ε, ως ευρωβουλευτές πρέπει βεβαίως να απευθυνόμαστε στους ψηφοφόρους μας και όταν υπάρχει βεβαίως κάποιος δημοσιογράφος ε, ε, και θέλει να πει κάτι για μας ή να δείξει κάποιο πλάνα καλό είναι να ακούγονται στην ε, γλώσσα μας οπότε είναι ως γνωστό έχουμε αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε 28 κράτη-μέλη αλλά πέρα από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών ε, οφείλω να πω, επειδή εγώ είμαι και από το Ολυμπούργο, πως υπάρχουν και μικρότερες ε, γλώσσες και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε τις ε, επίσημες γλώσσες παρά το ότι συχνά αυτές μιλούνται από μικρά ποσοστά των κατοίκων. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να μπορούμε να ειδοποιούμε και εμείς ως βουλευτές όταν δεν χρειαζόμαστε ε, την ε, διερμηνία. Ε, ο Ευρωπαίος φορολογούμενος αντιλαμβάνεται πως χρειαζόμαστε διερμηνής για να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά γεμάτες καμπίνες χωρίς βουλευτές από κάτω δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Ε, βεβαίως το κόστος ε, αντιστοιχεί σε 5 ευρώ αναπολίτη την ημέρα όπως ξέρετε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξοικονομήσεις με το να μοιράσουμε και εμείς καλύτερα τη δουλειά μας σε ολόκληρη την ε, εβδομάδα και βεβαίως ε, ωφελεί πάρα πολύ και το κόστος το να τελειώνουν ε, και πριν από τις 11 η ώρα το βράδυ οι συνεδριάσεις. Και στην εκθεσή μου αναφέρουμε ε, κάποια σημεία στα οποία θεωρούμε πως πρέπει να γίνουν κάποιες ε, βελτιώσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι, όπως είπαμε, τις πάρα πολύ καθυστερημένες ε, ακυρώσεις, οι οποίες ε, φτάνουν ένα 20% και μπορεί να κοστίσουν μέχρι και 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα κόστος το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται να πληρώνουμε και ε, ακριβώς το πληρώνουμε όταν δεν κάνουμε χρήση των υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να το γνωρίζουν το κόστος αυτό και οι βουλευτές πέρα από τους υπαλλήλους και τους βοηθούς. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, προτάσεις ε, κατόπιν ε, το, η διερμηνία on demand αναλόγως με τις ε, ε, γλώσσες οι οποίες απαιτούνται σε κάθε συνεδρίαση και βεβαίως θα πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη του κόστου το οποίο βεβαίως πρέπει να πω πως μειώνεται και να δούμε και το νέο γλωσσικό καθεστώς όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Κομισιόν το ε, Συμβούλιο και αλλού. Είχε γίνει μια σχετική μελέτη το 2005 αλλά πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά. Οπότε Αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουμε για την πολυγλωσία και τον περιορισμό του κόστους. Επίσης, ε, η απόφαση και η απέτηση που έχουμε και η βασική μας απέτηση είναι να υπάρξει μια απόφαση του Προεδρείου πριν από το τέλος του έτους. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ενθάρρυνση που μας δίνετε. Η κυρία Σπίκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θα ήθελα απλώ να διορθώσω κάτι. Είπατε 23 γλώσσες, 24 όμως είναι με τα κροατικά. Επίσης, θα συμφωνήσω με τις προτάσεις της έκθεσης ότι βεβαίως πρέπει να μειωθεί το κόστος. Υπάρχει το οικονομικό ε, επιχείρημα, το επιχείρημα της εξοικονόμησης. Όμως η γλώσσα μας σήμερα έχει μπει στις επίσημες γλώσσες. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να μιλήσουμε τη μητρική μας γλώσσα τα κροατικά. Ίσως κάποιοι δεν το παίρνουν τόσο σα σοβαρά, αλλά βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο για να γίνουν κάποιες εξοικονομήσεις, συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πολυγλωσία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε την πολυμορφία, την πολυγλωσία, συνεχίζοντας βεβαίως προσπάθειες για εξοικονόμηση. Σαν νέο μέλος επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μητρική μας γλώσσα. Ευχαριστώ. Κυρία εισηγήτρια, θεωρώ πραγματικά ότι πρόκειται για μία επιπλέον επίθεση κατά της πολυγλωσσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτήν την έκθεση, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του κόστους και της εξοικονόμησης, μειώνουμε το ποσό που διατίθεται για τη διερμηνία και μειώνονται οι υπηρεσίες οι οποίες ουσιαστικά στηρίζουν το δικαίωμα των βουλευτών να εργαστούν και να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αδυναμίες στην υπηρεσία διερμηνίας και μετάφρασης. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει διερμηνία σε κάποιες συνεδριάσεις προς και από όλες τις γλώσσες. Αυτές οι αδυναμίες δεν αρκούν για την εισηγήτρια. Θέλει κι άλλο ακόμα να πλήξει αυτή την υπηρεσία. Εμείς δεν πρόκειται να στηρίξουμε μια τέτοια επισφαλή κατάσταση, να την επιδεινώσουμε. Πρόκειται για παραβίαση των ε, δικαιωμάτων των βουλευτών να εργαστούν στη γλώσσα τους. Πρέπει να στηρίξουμε τους διερμηνείς και να υπάρχουν πολλοί άριθμοι στις συνεδριάσεις μας. Νομίζω όμως ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η συνεδρίαση στις 10 το πρωί, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί και το απόγευμα από τις 3. Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή νύχτα.